Ε, μαζί μου και από Λεμανία τη ε, στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο κύριος Λαμπρινίδης. Οι αρμόδιες ε, κυπριακές αρχές μου είπαν πως ο κύριος Σοφοκλής Σοφοκλέος καταλαμβάνει την θέση του κυρίου Κυριάκου Μαυρονικόλα από 1η Σεπτεμβρίου. Καλώς ορίζω τον νέο συνάδελφο και υπενθυμίζω πως σύμφωνα με τον κανονισμό απολαμβάνει πλήρη δικαιώματα και συμμετέχει στη συνεδριά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρκεί να έχει δηλώσει πως δεν κατέχει κανένα αξίωμα το οποίο είναι ασυμβίβαστο με αυτό του Ευρωβουλευτή. Οπότε κύριε Σοφουκλέους, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, ε, σύμφωνα με το άρθρο 3, στις 9 Ιουλίου εξέτασε τις εντολές των συναδέλφων Μπάνκι Μπάγκη από Ιουλίου 2009